Colleagues, if everyone is ready, we can begin. Do you want to take your seats? Everyone. Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. So, colleagues, this is a... Κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Πολιτικών Ελευθεριών, άρθρο 55. Χαίρομαι που έχουμε την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων μαζί μας για αυτή την κοινή ψηφοφορία για το πρόγραμμα για τα θέματα της δικαιοσύνης πριν προχωρήσουμε η Χάιντι Χάουλταλα από τη Τζούρι και ο κ. Βάιτερ Χόζερ από τη Λίμπε. Ένας από τους δύο θέλει να μιλήσει. Όχι, ψηφίζουμε λοιπόν. Έτοιμοι. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. ετοιμάστε τις κάρτες σας. Τροπολογία 101. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για τους συναδέλφους της Τζούρι. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 101. Έτοιμοι. Θα περιμένω ένα λεπτάκι για να καθίσετε ηρέμα, να μην τραυματιστείτε, να καθίσετε προσεκτικά. Ψηφίσατε όλοι. Συγγήτρια καταφθάνεια. Θα περιμένουμε μέχρι να ψηφίσει. Τι έγινε, πέρας. Όχι, ακόμα ανοιχτή ψηφοφορία. Okay, the rapporteur has voted. The co-rapporteur has voted. Ψηφίσανε λοιπόν. Πέρας. Jean can't cope with that long uh, delay really upset now. Το ταράξαμε το μηχάνημα και κόλλησε και είπα. Α, πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 122. Άρχεται. Η 122. Πέρας. Όχι μάλλον ακόμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3α. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 129. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 130. Άρχεται η ονομαστική κλίση. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 131. Άρχεται η νομαστική κλίση. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 132. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 133. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 134. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική πέντε. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 142. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Κόντ 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τοπολογία 6. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. 8 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. ΦΑΜ 29 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μπατζ 7 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τοπολογία 151. Άρχεται. Πέρας. Α, απορρίπτεται. Κόντ 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τοπολογία 152. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τοπολογία 153. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Α, απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. ΦΑΜ 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Άρχεται. Πέρας. Έγκρινεται. 55. Άρχεται. Πέρας. Έγκρινεται. Κον 4. Άρχεται η συμφορία. Πέρας. Έγκρινεται. Φάμε 7. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Κοντ 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. ΦΑΜ 8. Άρχεται. Πέρας. Έγκρινεται. Συμβιβαστική 15. Άρχεται. Πέρας. Έγκρινεται. Τροπολογία 61. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Ξεκινάμε. Τέλος. Εγκρίνεται. ΦΑΜ 10. Ξεκινάμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17 ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τοπολογία 70 υπέρ. Πέρας. Εγκρίνεται. ΦΑΜ 13 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 78. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Κοντ 10. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 21. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Την 79 θέλετε. Ζαμαρή. Την 79. Ζαμαρή. Ναι, 79. Ζητώ συγγνώμη. Δίκιο έχεις. Πάμε πίσω στην 79. Να ψηφίσουμε την 79 και θα κυρώσουμε τη συμβαστική 21 μέχρι να ψηφίσουμε την 79. Τροπολογία 79 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη συνάδελφοι. Συμβαστική 21 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23 άρχεται. Πέρας. Ε, εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 88. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Άρχεται. Α, συγγνώμη. ΦΑΜ 17. Άρχεται. Δεύτερο λάθος που κάνω. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Budget 2. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Budget 3. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 27. Άρχεται για τη συμβαστική 27. Πέρας. Εγκρίνεται. Τοπολογία 95. Ξεκινάμε. Α, όχι. Ναι, διότι αν είναι εγκριθεί, πάμε στην 95. 95. Πέρας. Πέρας. Εγκρινέται. Κοντ 15 άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται. Κοντ 16 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 28 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Μπότζε 4 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τοπολογία 11 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 99. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 29. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Budget 1. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 46 υπέρ, 6 ψήφια εναντίον, Δύο αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν στην κυρία Χάτολα και στον κύριο Βάιτεν Χόζα. Συγχαρητήρια συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τους συναδέλφους της Επιτροπής Τζούρι. No, we have more votes. We have more votes. So, um, Libe colleagues, if you could please stay and we begin our votes. Um... Συνάδελφοι της Λίμπε, μείνουν, ε, να ξεκινήσουμε τις ε, ψηφοφορίες. Ξαναξεκινάει το μηχάνημα. Δεν ξέρω τώρα πώς να πω στους συναδέλφους ε, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων να φεύγουν σιγά σιγά.